Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην καινούρια Επιτροπή Αναφορών, στην συντακτική της συνεδρίαση. Ονομάζομαι Κάρλος Ιτρουγκάη, του Λαϊκού Κόμματος ε, από την Ισπανία. Προεδρεύω αυτής της Επιτροπής, όχι επειδή είμαι ο πιο ηλικιωμένος ή ο παλαιότερος, αλλά γιατί αλλάζουν οι κανόνες και η γραμματεία μου ζήτησε να αναλάβω εγώ αυτό το καθήκον. Δεδομένου ότι ήμουν αντιπρόεδρος στην προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής. Έχουμε ανθρώπους πολύ παλαιότερους, όπως ο κύριος Κάσμαν, ο φίλος μου, που τα κατάφερε πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα θα μπορούσε να τα καταφέρει πολύ καλύτερα από μένα και σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει με χαρά μου ανέλαβα αυτή την υποχρέωση. Ας ξεκινήσουμε με την εκλογή της Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Για Πρόεδρο προτείνεται μία υποψηφιότητα η κυρία Ματσόνη του, της ομάδας του Λαϊκού Κόμματος. Υπάρχει κάποια άλλη μήπως υποψηφιότητα. Όχι. Ας κάνουμε την εκλογή διαβοής αν θέλετε υπέρ Δεχ χρειάζεται καν να πούμε ψήφι υπέρ. Το χειροκρότημα ήταν αρκετό, κυρία Ματσόνη. Θα ήθελα πολύ σύντομα να σας ευχαριστήσω όλους ε, διότι διαβοής με εκλέξατε στην θέση της Προέδρου. Ευελπιστώ ότι θα είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στις προσδοκίες όλων σας ε, και σε συνέχεια βεβαίως του έργου που ξεκίνησε η προηγούμενη Προεδρία πολύ γρήγορα τώρα προχωράω ε, στις υποχρεώσεις μου ως Προέδρου. Εδώ πρόκειται για την ε, συντακτική ε, συνεδρίαση και επομένως μπορούμε γρήγορα να προχωρήσουμε όπως γρήγορα πρέπει να προχωρήσει και η Ευρώπη. Εάν δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο, αλλά μάλλον είδα ότι κάποιος ήδη θέλει να ζητήσει το λόγο, και θα τον δώσω πριν εκλέξουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάσμαν λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα το λόγο για το επόμενο θέμα. Όταν θα το ανακοινώσετε λοιπόν τότε θα ξαναζητήσω το λόγο. Λοιπόν, για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου έχουμε μονάχα μία υποψηφιότητα. Αυτή είναι της κυρίας Παλιατέρη. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω διαβοής να εκλεγεί και η κυρία. Η κυρία Παλιαδέλη. Θα ήθελα να σας συγχαρώ βεβαίως, ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, η κυρία Παλιαδέλη δεν είναι εδώ. Α, εδώ είστε. ήθελα να πω εξ ονόματός της ότι δέχεται να είναι αντιπρόεδρος, αλλά ε, νομίζω ότι μπορεί να το πει η ίδια. Συγχαρητήρια λοιπόν κυρία Παλιαδέλη. Για την θέση του δεύτερου αντιπροέδρου έχουμε επίσης μία υποψηφιότητα μονάχα του κυρίου Μάγερ. Και προτείνω λοιπόν την ίδια μέθοδο διαβοής. Συγχαρητήρια και στον κύριο Μάγερ επί τη εκλογή του. Τρίτος αντιπρόεδρος. la Ωραία, ξανά έρχεστε λοιπόν, θαύμα. Ultima votazione per Τέταρτος αντιπρόεδρος. Χάνκης επίσης μοναδική υποψηφία. Quindi Επομένως, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους νεοεκλεγέντες αντιπροέδρους και βεβαίως να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Πρέπει να σας πω ότι πλέον έχει συσταθεί η Επιτροπή μας και ζητώ εάν κάποιος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, από την κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πήρα τον λόγο πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε το λόγο κυρία Πρόεδρε ε, και ζήτησα να μιλήσω για να πω δύο κουβέντες μόνο. Πρώτα απ' όλα το όνομα της Επιτροπής μας. Γνωρίζομαι ότι στην προηγούμενη θητεία είχε αναφερθεί ότι ο τίτλος της Επιτροπής θα πρέπει να αλλάξει, ας πούμε να γίνει Επιτροπή Αναφορών των ε, ε, Πολιτών σε ορισμένες ε, γλώσσες το όνομα της Επιτροπής μας ε, δεν είναι κατανοητό. Ας πούμε στα Δανέζικα που είναι η δικιά μου μητρική γλώσσα, ε, εάν ένας πολίτης της Δανίας ακούσει αυτήν την Επιτροπή δεν θα καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Θα πρέπει να την εξηγήσω λοιπόν εγώ κάθε φορά, πρέπει να εξηγώ στους πολίτες, στους συμπολίτες μου τι ακριβώς κάνει η Επιτροπή στην οποία συμμετέχω. Αυτή και περίφημη Επιτροπή Αναφορών. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από την νεοεκλεγήσα πρόεδρο και από τον νεοεκλεγέν προεδρείο να αρχίσουν τις συζητήσεις έτσι ώστε το όνομα, ο τίτλος της Επιτροπής να είναι κατανοητό από όλους τους πολίτες. Δεύτερον, Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να καλέσουμε την Σουηδική Προεδρία να έρθει στην Επιτροπή μας έτσι ώστε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να καλέσουμε την κυρία Σεσίλια Μάνστρομ, την ε, Υπουργό ε, για θέματα ε, με σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να έχουμε λοιπόν μία συνάντηση με την Προεδρεύουσα έτσι ώστε να ξεκινήσει μια στενότερη και καλύτερη συνεργασία ε, με το Συμβούλιο. Αυτά ήθελα να σας πω και νομίζω ότι καλό θα ήταν να έρθει η Σεσίλια Μάνστρομ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλα τα σημεία αυτά θα πρέπει να τα δούμε στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής ε, και βεβαίως ε, και αφού συναντηθούν και οι συντονιστές. Δεν νομίζω ότι πρέπει εδώ να ξεκινήσουμε τέτοια συζήτηση και βεβαίως να σας συγχαρώ και να σας πω ότι θα έχετε την πλήρη στήριξή μου κυρία Πρόεδρε. Øh, Μία ερώτηση ε, σχετικά με την ε, πρόσκληση ε, για τη Σουηδική Προεδρία. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε, αλλά καλά ήταν αυτό που είπατε σχετικά με το όνομα της Επιτροπής. Αυτό το έχουμε ήδη προτείνει, έχει αποφασιστεί από το Κοινοβούλιο. Άρα δηλαδή στην ιστοσελίδα, εκεί όπου παρουσιάζουμε το έργο μας. Ε, νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε και πόσο σημαντική είναι η Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και για μένα τα συγχαρητήριά μου και από μένα τα συγχαρητήριά μου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πραγματικά έχουμε την ευκαιρία σε αυτήν την Επιτροπή με τη Σουηδική Προεδρία να εισάγουμε ένα νέο πολιτισμό, μια νέα νοοτροπία. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε από το Συμβούλιο ότι όταν υπάρχουν αναφορές συγκεκριμένων κρατών μελών θα πρέπει να έρχονται πιο συχνά οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου. Αυτή είναι μια πρόταση που νομίζω μπορούμε να τη θέσουμε άμεσα στους συντονιστές. Τώρα, όσον αφορά τις αναφορές, το petition έρχεται από μια λατινική λέξη. Ε, οι Γερμανοί παρότι χρησιμοποιούν άλλες ε, λέξεις ε, καταλήγουν στη λέξη ombudsman. Αν λοιπόν βάλουμε στα γερμανικά τουλάχιστον αντί για petition σε τη γερμανική λέξη του πολίτη τα πράγματα θα γίνουν πιο μπερδεμένα. Εν πάση εγώ θεωρώ ότι η Επιτροπή αυτή έχει μία ονομασία που είναι καταχωρημένη. Δεν πρέπει λοιπόν να βιαστούμε να αποφασίσουμε. ω εκ τούτου θα πρέπει να περιμένουμε μία πρόταση από το Προεδρείο του τι θα κάνουμε στο μέλλον. Και να θίξω κάτι όπου κατά την άποψή μου θα ήταν σημαντικό. Δεν ξέρω αν την επόμενη εβδομάδα θα είσαστε στις Βρυξέλλες, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά ε, το Προεδρείο να συνεργαστεί με τη Γραμματεία ταχύτατα. Έχουμε πολλές αναφορές που εκκρεμούν εδώ και χρόνια και όπου οι πολίτες έχουν απογοητευτεί. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν κάποιες ε, αναφορές να τις ε, επιταχύνουμε και έχουμε συγκεκριμένα έχω κατά νου μία αναφορά όπου μας ε, έχουν προσκαλέσει να επισκεφθούμε μία ορεινή περιοχή για να δούμε ζημιές που έχουν προκληθεί. Ίσως αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε το καλοκαίρι, αλλά από το Σεπτέμβρη. Αν όμως ε, περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβρη, τότε πλέον οι ζημιές δεν θα είναι ορατές ε, λόγω του χιονιού ε, και θα έχουμε χάσει την ευκαιρία, δηλαδή κρίμα η αναφορά. Πρέπει ως εκ τούτου να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούμε να περιμένουμε να περνάνε δύο μήνες. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι θαυμάσιο το ότι στο Προεδρείο τουλάχιστον επιτέλους ε, έχουμε κάποιο αντίβαρο περισσότερες γυναίκες. Όπως ξέρετε το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία, καλύτερα να μην μιλάμε πολύ. Εγώ προτείνω λοιπόν οι δύο προτάσεις που σας έχουν κατεθεί, η πρόσκληση της Σουδικής Προεδρίας και η αλλαγή της ονομασίας επιτροπής να μην βιαστούμε. Δεν πρέπει, συνήθως συμφωνώ με την προελίσσα, αλλά εδώ λέω να μην βιαστούμε να συναντηθούν οι συντονιστέ με το Προεδρείο και μετά να καταλήξουν σε μια λογική απόφαση την επόμενη φορά, όποτε και αν είναι αυτή. Ε, αυτό έχω να σα προτείνω, ε, κύριε Πρόεδρε. Sí, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ και την Πρόεδρο και τους και τις Αντιπρόεδρους. Σε αυτή την Επιτροπή έχουμε πλέον ε, περισσότερες γυναίκες από ότι άντρες. Αλλά να πω το εξής, το όνομα μιας Επιτροπής δεν το αποφασίζει η ίδια η Επιτροπή. Δεν είμαστε σε ένα Σοβιέτ ε, που αποφασίζει ω αυτόνομο όργανο. Αν θέλουμε μπορούμε να ζητήσουμε αλλαγή ονόματος, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία γι' αυτό. Αν επιθυμούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, να το κάνουμε. Αλλά σίγουρα δεν έχει αυτό το δικαίωμα κάθε επιτροπή. Δηλαδή, φανταστείτε την Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων ή την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ξαφνικά να βγει και να αλλάξει το όνομά τη τα ονόματα αποτελούν ε, τμήμα του, στη συνολική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Συνεπώ, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαδικασία πρόταση ενό καινούριου ονόματο. Αλλά αυτό δεν είναι ε, δική μας ε, δουλειά και ιδιαίτερα όχι σήμερα. Συμφωνώ να το αναβάλουμε, όπω είπε ο κ. Κάσμαν. Θα ήθελα όμω να σα πω ότι αυτό έχει ήδη αποφασιστεί. Πολλοί από εσά είστε καινούργοι, αλλά είχε αποφασιστεί από το, το προηγούμενο κοινοβούλιο, από την προηγούμενη σύνθεση. Δεν είναι κάτι καινούργιο, έτσι. Δεν το βγάζω εγώ από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Η αλλαγή του όνομα τη είχε ήδη αποφασιστεί. Δεν τη βγάζω εγώ από το καπέλο μου. Συμφωνώ όμω να αναβάλουμε την απόφαση γιατί είναι πολύ σημαντική απόφαση. Θα μπορούσε να βοηθήσει ορισμένου από εμά, λίγου ίσω, αλλά θα μα βοηθούσε πολύ. Ωραία, θα, περά... θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο, ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα, είναι έμπειρος. Ακούσαμε τους συναδέλφους και σήμερα στην μερίσια διαταξή δεν προβλέπεται καν αυτό το θέμα. Οπότε προτείνω να το συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση συντονιστών. Γιατί σήμερα η συνάντηση είναι συντακτική αυτή η συνεδρίαση. Κυρία Άουκεν, θα είμαστε πολύ καιρό μαζί, θα μάθουμε πολύ καλά ο ένας τον άλλο και θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Πολύ ωραία. Ε, συμφωνώ με τον Αντιπρόεδρο. Και άλλωστε αυτό θα είχα προτείνει και εγώ η ίδια. Είχα σκεφτεί δηλαδή να ε, συγκληθεί η συνεδρία των συντονιστών για την 26η Αυγούστου έτσι ώστε ε, να προετοιμαστούμε για την 1η Σεπτεμβρίου οπότε θα λάβει χώρα και η πρώτη συνάντηση συνεδρίαση της Επιτροπής ε, και νομίζω ότι τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία εθίγησαν μόλις τώρα και βεβαίως να συζητήσουμε και το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της Επιτροπής ε, ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη στήριξη από τους ε, πολίτες της Ευρώπης το δε ενδεχόμενο της πρόσκλησης εκπροσώπου της προεδρεύουσας χώρας, της Σουηδίας, βεβαίως είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρότασης γιατί μας ενδιαφέρει να υπάρχει καλή και εντατική συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα θεσμικά όργανα έτσι ώστε να μικρύνει όσο γίνεται περισσότερο ο χρόνος αντιμετώπισης αυτών των ε, καταγγελιών που φτάνουν στα χέρια μας από πλευράς των ε, πολιτών. Και βεβαίω, όπω έλεγα και προηγουμένω, να συνηθούν πρώτα οι συντονιστέ να παίξουν το σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να παίξουν σε όλη τη διάρκεια τη επόμενη θητεία ε, και επομένω ε, κλείνοντας να συγχαρώ όλους τους νεοεκλεγέντε, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τη Επιτροπής και θα συναντηθούμε τέλη Αυγούστου.